την πρόταση για τους διορισμούς για τη σύνθεση των ε, επιτροπών. Οι προτάσεις δημοσιεύτηκαν στις, ε, στην ενημέρωση της, ε, για την Ολομέλεια στο site της, του Κοινοβουλίου και μέχρι αύριο στις 10 μπορεί να καταθέσετε